Ελπίζω να ξεκουραστήκατε όλοι στις ε, διακοπές και σίγουρα άλλαξαν πολλά πράγματα σε σχέση με το παρελθόν ε, για τις ε, διακοπές μας. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και με στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ήμουν σε διαρκή επαφή με την Πολωνία.